So, dear colleagues, let's start. Unfortunately, we are a little bit late because uh, we had this common meeting. Ας ξεκινήσουμε, συνάδελφοι, γιατί είχαμε αυτήν την ε, κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή ΑΦΕΤ. Και όπως γνωρίζετε βέβαια, πολύ μακρηγορούν στην Επιτροπή ΑΦΕΤ, οπότε χρειαστήκαμε λίγο παραπάνω χρόνο. Λοιπόν, περνάμε στο σημείο 2 της σημερινής σας διάταξής μας. Έγκριση της σημερινής σας διάταξης έλαβα από μια σειρά από πολιτικές ομάδες ε, ένα αίτημα για προσθήκη στην ημερήσια διάταξη σε ό,τι αφορά μια προφορική ερώτηση σε σχέση με την Ορβηγία και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, θα σα πρότεινα να εγκρίνουμε με αυτή την προσθήκη την ημερήσια διάταξη. Καλώς λοιπόν. Σημείο 3. Ανακοινώσει του Προέδρου. Καταρχήν θα ήθελα να σα ενημερώσω για μία ακόμα φορά ότι Έχουμε web streaming αυτή τη συνεδρία σήμερα, οπότε καλωσορίζουμε και όλους όσους μας παρακολουθούν εκτός Βρυξελών και καλό είναι να το έχετε αυτό κατά νου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής μας. Από εκεί και μετά ενημερωτικά σε ό,τι αφορά τη μακροοικονομική υποστήριξη προς την Ουκρανία να πούμε πως η δεύτερη δόση έχει πλέον αποδεσμευτεί έτσι ώστε η Ουκρανία από το 2014 να έχει λάβει 2,81 δις ευρώ. Αναφερόμαστε δηλαδή ε, για το μεγαλύτερο ποσό στο πλαίσιο μακροοικονομικής υποστήριξης που έχει παράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν υιοθετήθηκε το σχετικό πρόγραμμα MFI και από εκεί και μετά στις Ηνωμένε Πολιτείες τώρα έχουμε τη διαδικασία του διορισμού του USTR, του κυρίου Ρόμπερτ Λάιτχαζ, του οποίου η ακρόαση στο Κογκρέσο και, στο, και στη Γερουσία έγινε ήδη, αλλά ενδεχομένω να υπάρξουν κάποια διαδικαστικά ζητήματα ακόμα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν μέχρι να αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του. Ίσως δηλαδή να περάσουν μερικές εβδομάδες ακόμα μέχρι να αναλάβει. αλλά από εκεί και μετά έχουμε κύριο Ναβάνου, κύριο Μος, ως Υπουργό Εμπορίου και ως γεωστιάτο τον κύριο Λάιτ Χάζερ, οπότε έχουμε τα τρία αυτά άτομα με κεντρικούς ρόλους σε ό,τι αφορά την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ, σε ό,τι αφορά τη χώρα την, ε, την Αζία. Βλέπουμε πως ε, έχει τεθεί και πάλι επιτάπητος ε, το ζήτημα σύναψης μια εμπορική συμφωνία με την Αζία. Όπως θα θυμόσαστε είχαμε ξεκινήσει τις σχετικές διαπραγματεύσεις το 2007 και υπάρχει μια εντολή για σύναψη συμφωνίας με την Αζία. Ωστόσο, στο ενδιάμεσο διάστημα είχαμε τη δυνατότητα να προβούμε σε διμερείς διαπραγματεύσεις με μια σειρά από χώρες της Αζία. Ωστόσο τώρα ε, η κατάσταση έχει αλλάξει λίγο γιατί τον ε, Μάρτιο η Επίτροπο ε, Μάρτιο ε, συναντήθηκε με του αρμόδιους υπουργού των χωρών τη ΑΣΕΝ και θεωρείται ότι μπορούν να ξαναρχίσουν οι σχετικές προπαρασκευαστικές εργασίες για την σύναψη μιας συμφωνίας με την Άζια, γεγονό το οποίο είναι θετικό. Τώρα, σημείο 4, το οποίο αφορά και ένα νέο σημείο εδώ στην Μέση αφορά τις, ε, τη νέα διαδικασία που προβλέπεται εδώ για τις συνεδριάσεις μας και η οποία συνεπάγεται ότι θα πρέπει να διαβάζετε πολύ προσεκτικά τα όσα, τις ε, σημειώσεις σε σχέση με τις αποφάσεις που λαμβάνονται στις ε, συνεδριάσεις των συντονιστών, όπως δημοσιεύονται. Ούτω ή άλλω αυτό γινόταν καθέν, αλλά τώρα καλούμαστε λοιπόν με βάση την εμερήσια διάταξή μα να εγκρίνουμε αυτέ τι αποφάσει που λαμβάνονται από, την, από τους συντονιστές συνεδρίασή τους. Οπότε αυτός ε, που σας προτείνω είναι να δούμε ποιες ήταν οι αποφάσεις που ελήφθηκαν η τελευταία συνεδρίαση της, ε, των συντονιστών στις 27 δηλαδή Φεβρουαρίου και αν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις μέχρι την ολοκλήρωση τη σημερινή μα συνεδρίασης, θα θεωρήσουμε ότι έχουν εγκριθεί εν λόγω αποφάσει. Σε διαφορετική περίπτωση, προφανώ θα τη συζητήσουμε. Περνάμε στο σημείο 5. Και αυτό το σημείο εδώ λοιπόν αφορά την ε, Ουκρανία και την υποστήριξη που έχουμε παράσει προς αυτή τη χώρα. Και εδώ αναφερόμαστε σε πιο συγκεκριμένα σε προσωρινά αυτόνομα εμπορικά μέτρα για την Ουκρανία. Νομίζω πως ε, και αυτά τα εμπορικά μέτρα αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης της Ουκρανίας. 65 τροπολογίες έχουν κατατεθεί από μέλη εδώ της ΙΝΤΑ και από εκεί και μετά έχουμε και την ομοθέτηση από την πλευρά της ε, Επιτροπής Άγκρη. Να δώσω όμως το λόγο στον ε, Συγχαρητή τον κύριο Βαλέση. Να τους ευχαριστήσω όλους για την συνεισφορά τους στο σχέδιο έκθεσης. Θα ξεκινήσουμε με τις τροπολογίες στην πρόταση της Κομισιόν και μετά θα περάσω στα παραρτήματα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα των διασφαλίσεων. Φαίνεται ότι οι βουλευτές συμφωνούν ότι χρειαζόμαστε έναν ισχυρότερο τέτοιο μηχανισμό, όμως υπάρχει διαφορετική άποψη για το πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Για εμένα ήταν σαφές εξ αρχής ότι ο στόχος ε, των, της διαδικασίας αυτής είναι να μπορέσει η ευρωπαϊκή βιομηχανία να προστατευτεί από εισαγωγές και θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει τέτοιες δράσεις. Δεν υπάρχει νόημα να έχουμε τέτοια διαδικασία, δεν μπορεί να την ξεκινήσει η βιομηχανία. Επίσης, πρέπει να αποφασίσουμε ποιον ορισμό της βιομηχανίας θα χρησιμοποιήσουμε. Στο σχέδιο χρησιμοποίησα αυτόν που υπάρχει στην ε, Συμφωνία Ελευθερία με την Κορέα, που είναι ο πιο σύγχρονος. Και αυτή τη στιγμή συγκριθεί, δεν νομίζω ότι υπάρχει νόημα να δοθεί τέτοιο δικαίωμα στο Κοινοβούλιο, γιατί απλά θα καθυστερήσει η διαδικασία. Δεύτερον, κάποιε αυτοτροπολογίε έχουν εμπνευστεί από το μηχανισμό σταθεροποίηση τη μπανάνα, που ίσω δεν είναι ότι το καλύτερο, γιατί η κατάσταση είναι τελείω διαφορετική. Ο μηχανισμό αυτό είναι ένα μηχανισμό που βασίζεται σε κάποιο κατόφλι και έτσι έχουμε κάποιους μη προτιμησιακούς ε, δασμούς ε, που μπορεί να επανεισαχθούν μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους ε, μόλις φτάσουμε ένα κατόφλι. Στην περίπτωση της Ουκρανίας οι προτιμήσεις είναι υπό μορφήν ποσόστοσης χωρίς δασμούς, ε, παραδείγματο χάρη ε, υπάρχουν μη προτιμησιακή απλαγή από δασμούς ε, και οι δασμοί επιβάλλονται όταν φτάσουμε το ποσόστοση. Επίσης, εξαντούνται σε λίγες ημέρες. Οπότε, ο μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης επίσης δεν λειτουργεί. Συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει στενή παρακολούθηση της επίδρασής του στην αγορά, δεδομένου του ότι δεν έγινε κάποια αξιολόγηση αντικτύπου, όπως το 2007 όταν διαπραγματευτήκαμε την συμφωνία. Θα προτείνω κάποιες συμβαστικές τροπολογίες και κάποιες από τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί άλλαξαν την διατύπωση σε συνεχή παρακολούθηση που είναι κάτι το διαφορετικό. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω και μια συμβαστική λύση για τα παραρτήματα και αν δεν είναι αρκετά γενναιόδωρο δεν έχει νόημα να ζητάμε από την Κομισιό να κάνει αιτήσει ή μεσοπρόθεσμες ε, αναθεωρήσεις. Επίσης θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την διαφθορά πράγματι και πρέπει να το αναφέρουμε στο έγγραφο επιπλέον. Κάποιες από τις ε, τροπολογίες εξετάζονται από πλευράς διατύπωσης για το πώς οι διατυπώσεις αυτές είναι ε, από τη σκοπιά της συνεκτικότητας και της τυποποίησης των νομικών εγγράφων και θα επανέλθω σε αυτό και θα προτείνω κάποιες αλλαγές. στην συνεδρία των σκηνοδών. Περνάμε τώρα στις ε, τροπολογίες, ε, στις τροποποίησεις των παραρτημάτων. Πριν από μια εβδομάδα η Επιτροπή Άγκρη ψήφισε και τα μέλη της Επιτροπής αποφάσισαν να διαγράψουν τις γραμμές για σε καλαμπόκι, στάρι, κρυθάρι, επεξεργασμένες ντομάτες από τις 55.000 50.000 τόνους και στην Επιτροπή ΙΝΤΑ έχουμε τροπολογίες που ζητάνε να διαγραφούν σχεδόν όλες οι δασμολογικές γραμμές γεωργικών προϊόντων και να αυξηθούν οι ποσότητες προτείνει η Κομισιόν. Συνεργάζομαι εδώ με τους συναδέλφους για να καταλήξουμε σε κάποιες συμβιβαστικές προτάσεις για τα γεωργικά προϊόντα. Ήδη την προσωπική μου άποψη την έχω εκφράσει. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια διαφοροποίηση των εξαγωγών και να στηρίζουμε με τις συμφωνίες αυτές τις μικρομεσαίες Υπήρχαν τροπολογίες που διέγραφαν την ουρία για λείπασμα είναι ένα ευαίσθητο προϊόν στην βιομηχανία, ιδιαίτερα ευπαθές, καθώ έχει, έχουν υπάρξει μία ανταγωνιστικές πρακτικές στο παρελθόν και η Κομισιόν αντέδρασε επιβάλλοντας δασμούς αντι-dumping για προϊόντα που εξάγει η Αλγερία, η Λευκορωσία, Ρωσία και η Ουκρανία και συμφωνώ με τους συντάκτες ε, των τροπολογιών αυτών για να διαγραφεί το λείπασμα αυτό. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι αντιλαμβάνομαι την μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ουκρανία. Πολεμάει έναν εξωτερικό εχθρό και ταυτόχρονα πρέπει να κάνει μεταρρυθμίσεις. Γνωρίζω ότι και το εμπάργο και η απαγορευσή διέλευσης έχει επηρεάσει πολύ το εμπόριο και πρέπει να το έχουμε και αυτό κατά νου. Τέλος, πρέπει να αναφερθώ σε κάτι σημαντικό. Την απαγόρευση εξαγωγής ξυλίας. Παρατηρούμε τις εξελίξεις στην ομοθεσία και ελπίζω ότι θα υπάρξει σχετική νομοθεσία. Αλλά η απαγόρευση αυτή είναι κατά των κανόνων του ΠΟΕ και των ε, Κανόν της ε, Συμφωνίας του Βορείου. Πρέπει να το έχουμε κατά νου αυτό. Και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πίεση βεβαίω, αλλά να το ξαναπώ. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Πρέπει να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Σας ευχαριστώ. Οι οι συγητές για τους σοσιαλδημοκράτες, η Μαρίτα Ολφσκόπ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 Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε. Ήδη πολλάκις είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα της βοήθειας για την Ουκρανία φορά και το θέμα που συζητάμε σήμερα. Θα ήθελα λοιπόν να υπενθυμίσω στην εσωτερική αρχή μας εδώ πέρα ότι επιθυμούμε μια σταθεροποίηση της οικονομικής κατάστασης στην Ουκρανία, την οποία σημειώνουμε. Ταυτόχρονα όμως θέλουμε να επιμείνουμε στο μηχανισμό παρακολούθησης έτσι ώστε όλοι οι όροι που υπάρχουν ε, να τηρηθούν ελπίζοντας ότι θα οδηγηθούμε σε μια πραγματική αλλαγή της ε, ακόμα μη ικανοποιητική κατάστασης όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ουκρανία. Και θα ήθελα άρα να υπενθυμίσω τις τροπολογίες 2 και 4 που ξεκαθαρίζουν ακόμη μια φορά πως ε, η αρισιμότητα αυτή πρέπει να διατηρηθεί σε όλη την διαδικασία της παρακολούθησης. Δηλαδή, σε περίπτωση που δεν εκπληρωθούν αυτοί οι όροι από την ε, Ουκρανία και έχουμε επαναφορά των πληρωμών, κάτι το οποίο θα είναι νομίζω μια προϋπόθεση για την θετική κατάληξη όλων αυτών των εμπορικών μέτρων για την εμπορική συνεργασία δηλαδή και θεωρώ πως η Κομισιόν θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική και να φροντίζει να εκτιμά το κάθε έτος ε, που περνάει ακριβώς και να ενημερώνει το Κοινοβούλιο για τα μέτρα για να μπορούμε και εμείς να αποφασίζουμε υπεύθυνα το τι θα κάνουμε. Οπότε... Αναμένω βεβαίως και την επικοδομητική συνεργασία με τους υπόλοιπους ε, σκιώδεις εισηγητές. Σας ευχαριστώ. Χάιντι τη Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Η Ουκρανία εξαρτάται εντυπωσιακά από τη Γεωργία. Οπότε, εάν θέλουμε να βοηθήσουμε τη χώρα, δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε όσον αφορά το να βάλουμε στην άκρη το σύτο και το καλαμπόκι όσον αφορά αυτά τα μέτρα. Να μην είναι αυτή η γραμμή μας. Και θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημοσιεύσει την αξιολόγηση. Έχουμε μια σχετική τροπολογία και άλλη μία που λέμε ότι για να μην έχουμε ε, ανανέωση των αυτονόμων εμπορικών μέτρων θα πρέπει να έχει προηγηθεί μια μελέτη επιπτώσεων. σύμφωνα και με συνέδελφο που είπε ότι θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο τις μεταρρυθμίσεις. Και σχετικά με τη διαφθορά. Μιλάμε στην ε, τρίτη μας τροπολογία. Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση της χώρας θα πρέπει αυτό να το θεωρήσει ως αντάλλαγμα αυτών των εμπορικών μέτρων. Ο Πρόεδρος. Ο λόγος τώρα στην Επιτροπή. Δεν ξέρω ποιος την εκπροσωπεί σήμερα. Καλησπέρα. Θα ήθελα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να σας ευχαριστήσω για το έργο που έχετε καταβάλει μέχρι τώρα και για τη συνεργασία που είχαμε. Γιατί προσπαθούμε βέβαια ε, και εμεί ε, να σας δίνουμε όσο περισσότερες πληροφορίες για τη σχέση με αυτό το ζήτημα. Θα ήθελα τώρα να θίξω μια σειρά από ζητήματα που τέθηκαν στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης. Ε, καταρχήν ε, διαπίστωσα ότι οι μέλη εδώ ε, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου θέλουν να υπάρχει μια όσο το δυνατόν πιο ισχυρή ρήτρα διασφάλιση, η οποία θα προστατεύει την αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγματι, αυτό είναι κάτι που επιθυμούμε και εμεί από την πλευρά τη Επιτροπή και θα πρέπει λοιπόν να βρούμε την κατάλληλη διατύπωση αυτή τη ρήτρα διασφάλιση, όπως θα περιλαμβάνεται στη δική μα πρόταση. για παράδειγμα, η διερεύνηση θα μπορεί να γίνεται μετά από σχετικό αίτημα ενό ε, κράτου μέλου, είτε μετά από σχετικό αίτημα ε, μιας, ε, ενός φορέα με νομική προσωπικότητα ή από την πλευρά μιας ένωσης πολιτών. Οπότε ενδεχομένω και πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να βρούμε μια καλή λύση συμβιβασμού σε ό,τι αφορά τώρα την παρακολούθηση, το ε, monitoring, διαπιστώνουμε ότι με βάση τις ε, τροπολογίες ε, που έχουν κατατεθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καλείται να παρακολουθεί την εφαρμογή των, του κανονισμού σε ό,τι αφορά τα ATMs, τα αυτόνομα εμπορικά μέτρα, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι Ούτω ή άλλω, εμεί από την πλευρά τη ε, Επιτροπή παρακολουθούμε το τι σημαίνει σε σχέση με τι δασμολογικέ ποσοστώσει, ε, τα TRQ. Και αυτό συμβαίνει και, ε, δηλαδή, παρακολούθηση από την πλευρά τη Επιτροπή και σε ό,τι αφορά τι τιμέ των αγροτικών προϊόντων, τι οποίε δηλαδή προβαίνει στην δημοσίευση τακτικών εκθέσεων η Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την τακτική υποβολή εκθέσεων, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των αυτόνομων εμπορικών μέτρων, να σα πούμε ότι θα υπάρξει ετήσια έκθεση από τη δική μας πλευρά και η πρώτη από αυτές τις εκθέσεις θα υποβληθεί φέτος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε, ναι, μπορούμε να σας να δεσμευτούμε ότι θα υπάρχουν εκθέσεις από την πλευρά σε ό,τι αφορά τα στατιστικά στοιχεία, σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές, αλλά ε, και τις δασμολογικές ποσοστώσεις. Κάτι τέτοιο δηλαδή είναι αυτονόητο ότι θα περιλαμβάνεται στην έκθεση. Αλλά επιτρέψτε μου να σχολιάσω ένα ζήτημα. Και αυτό είναι το εξή. Εάν μέσω της παρακολούθησης είμαστε σε θέση να ταυτοποιήσουμε ε, τους επιμέρους εξαγωγείς οι οποίοι αποφελούνται από αυτά τα αυτόνομα εμπορικά μέτρα, τότε ε, κάτι τέτοιο δεν θα είναι δυνατόν. Δηλαδή, το σύστημα διαχείρισης των, των δασμολογικών προσωστώσεων που χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή βασίζεται ε, στην αρχή του ο πρώτος ο οποίος ενδιαφέρεται είναι εκείνος που λαμβάνει ε, την ε, ποσότητα σε ό,τι αφορά δηλαδή την, την ποσότητα η οποία χορηγείται στον κάθε ε, και τη σχετική αδειοδότηση. Έτσι λοιπόν, ε, όπως είναι διαμορφωμένο αυτό το σύστημα διαχείρισης, δεν επιτρέπει την ταυτοποίηση συγκεκριμένων εξαγωγείων... οι οποίοι εποφελούνται από αυτά τα μέτρα για λόγους απορρίτου και για λόγους ενδεχόμενης σύγκρουση συμφερόντων. Οπότε τέτοιου είδους στοιχεία σε ό,τι αφορά μεμονωμένους εξαγωγείς δεν θα σας διατεθούν στο πλαίσιο της ε, παρακολούθησης του monitoring από την πλευρά της Επιτροπής. Ωστόσο, θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι εκείνες που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων οι οποίε δραστηριοποιούνται και δημιουργούν θέσεις εργασίας στον αγροτικό τομέα της Ουκρανίας, σύμφωνα με ανεξάρτητες μελέτε, συμπεριλαμβανομένε και τις μελέτες σε ό,τι αφορά ε, την ε, αξιολόγηση αντικτύπου του 2016. Άρα λοιπόν με βάση τα στοιχεία που έχουμε εμείς στη διάθεσή μας, το 75% της παραγωγής ε, ε, προέρχεται ακριβώς από αγροτικά νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες και απασχολούν το 90% του εργοτικού δυναμικού στον γεωργικό τομέα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό χωρίς βέβαια να αρνούμαστε την ύπαρξη πολύ μεγάλων επιχειρήσεων, ε, εμπορικών επιχειρήσεων στον ακροτικό τομέα, θα πρέπει να πούμε ότι τέτοιου είδους μέτρα στον ε, ακροτικό τομέα πραγματικά μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην αύξηση των εσόδων, ειδικότερα δε στον ε, κλάδο των δημητριακών, όπως αναφέρθηκε η σχετική έκθεση ΕΣΑΕ το 2007. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά και τα σχετικά μέτρα, θεωρούμε πως ε, αυτά τα μέτρα θα έχουν ιδιαίτερο αντίκτυπο στις υπεύθυνε αγροτικές ε, περιοχές ε, της Ουκρανίας. Και αυτό είναι σημαντικό να το γνωρίζετε στο πλαίσιο των συζητήσεων που θα κάνετε σε ό,τι αφορά τα προϊόντα, προϊόντα συγγνώμη, τα οποία θα περιληφθούν στα αυτόνομα εμπορικά μέτρα. Και εμείς ανησυχούμε ιδιαίτερα με τι ε, απόπειρε ε, που γίνονται για τον αποκλεισμό ορισμένων κατηγοριών ε, προϊόντων από την πρόταση. Γιατί όταν διαβάζουμε κάποιες από αυτέ τροπολογίε που έχουν κατατεθεί, σε ό,τι αφορά αυτά τα προϊόντα, διαπιστώνουμε ότι το 98% του συνόλου των εισαγωγών που δικαιούνται ATM θα αποκλείονταν από το πεδίο εφαρμογής τη ειδική πρόταση. Ουσιαστικά δηλαδή θα έχανε κάθε νόημα η πρόταση αν δεχόμασταν ε, την εξαίρεση αυτών των κατηγοριών προϊόντων. Οπότε θα ήθελα να σας, καλέσω, σας παρακαλέσω μόνο θερμά να επανεξετάσετε αυτές τις προτάσεις γιατί τα εν λόγω προϊόντα δεν αποτελούν κίνδυνο για την ε, αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν ε, ρίξουμε μια ματιά και στα σχετικά δεδομένα για το 2016, θα διαπιστώσουμε ότι οι εισαγωγέ από την Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση των εν λόγω προϊόντων, των περισσότερων από αυτά τα προϊόντα, ουσιαστικά μειώθηκαν. Και αυτό βέβαια συνηγορεί προς την πρόταση που έκανε η Επιτροπή το Σεπτέμβριο του 2016 η Επιτροπή. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ένα συμπληρωματικό ερώτημα από τον κύριο Σόλτς. Ναι, θα ήθελα ε, αφού άκουσα την Επιτροπή να θέσω ένα ερώτημα προς αυτή. Όταν μας λέτε ότι δεν είστε σε θέση με βάση την τρέχουσα μεθοδολογία σας για την παρακολούθηση να ε, γνωρίζετε το τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν θα πρέπει να αλλάξει αυτή η μεθοδολογία. Δηλαδή δεν θα πρέπει να γνωρίζετε ε, ποια είναι τα μερίδια της αγοράς και σε ποιον ανήκουν. Και αν δούμε για παράδειγμα της, ε, τον, ε, τον τομέα αυτών των εξαγωγών, ουσιαστικά έχουμε δύο κύριε επιχειρήσει εξαγωγών οι οποίε ελέγχουν το σύνολο τη αγορά τη Ουκρανία. Και οι οποίε δηλαδή ουσιαστικά ελέγχουν όλη την εξαγωγική ροή, τι εξαγωγικέ ροέ προϊόντων από την Ουκρανία προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, ε, πώ ε, θεωρείτε ότι θα αποφεληθούν κυρίω οι μικρομεσαίε επιχειρήσει Δηλαδή πραγματικά θα πρέπει να δούμε ποιος είναι τελικά εκείνος ο οποίος επωφελείται σε τελική ανάλυση από αυτά τα αυτόνομα εμπορικά μέτρα και κατά πόσο δηλαδή αποβαίνουν προς όφελος και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της ανάπτυξης της βιωσιμότητας. Και βέβαια και κατά πόσο και το όφελος ε, είναι υπαρκτό, είναι αυτό και ε, για τις ε, επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες για όλα αυτά τα ζητήματα σε διαφορετική περίπτωση ε, ε, προκύπτουν αυτά τα ζητήματα, όπω για παράδειγμα αυτά που αναφέρατε σχέση με τι τροπολογίε από την Επιτροπή Άγκρη, οι οποίε προτείνουν εξαίρεση κατηγοριών προϊόντων που καθιστούν άκυρη την πρόταση. Η Επιτροπή. Ναι, ε, σα είπα ότι υπάρχουν μεγάλε εξαγωγικέ επιχειρήσει που δραστηριοποιούνται στην αγορά, αλλά σα σας είπα επίση ότι μέσω τη δημιουργία νέων ευκαιριών για δραστηριοποίηση στην αγορά, ακριβώ επιτρέπουμε και την ενεργοποίηση ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όταν αναφερόμουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, έκανα λόγο για μικροπαραγωγούς, για οικογενειακές επιχειρήσεις. Ε, δεν αναφέρομαι δηλαδή στους, στους εμπορευόμενους. Εδώ αναφερόμουν στους παραγωγούς, γιατί δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με εμπορικές επιχειρήσεις αλλά και ε, παραγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει να επωφεληθούν έστω και έμεσα από την πρότασή μας αφού ε, με τις προτάσεις δημιουργούμε δυνατότητε ε, αύξησης της παραγωγής δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τονώνουμε την ανάπτυξη στις περιοχές εκείνες της Ουκρανίας οι οποίε ακριβώ θα υποφεληθούν από την πρότασή μα. Ευχαριστώ ο μας, ο κύριος Βαλέσα. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε τις μεταρρυθμίσεις ε, στην Ουκρανία. Τούτου λεχθέντος πρέπει στην Επιτροπή μας ε, να αναρωτηθούμε το εξής. Πρέπει να αγνοήσουμε την πρόταση των συναδέλφων της Επιτροπής ε, Γεωργίας. Πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Θα συναντηθούν οι σκιώδεις την Δευτέρα στις 4 η ώρα, οπότε μέχρι τότε θα σας παρουσιάσω την πρότασή μου για το πώς ε, θα έχουμε και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Σας ευχαριστώ. Η ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για τις 4 Μαΐου. Τελειώσαμε με το θέμα 5 και περνάμε στο 6. Το θέμα της εμπορικής πολιτικής και της ε, παγκοσμίας ε, αλυσίδας αξίας. Στο 70% του εμπορίου συνδέεται με αυτό. Και ε, έχουμε και το έγγραφο εργασίας από την εισηγήτρια την κυρία Αρένα και θα της δώσω τον λόγο. Πάρα πολύ θετικό το ότι αποφάσισε η Επιτροπή μα να φτιάξει αυτή την έκθεση. Γιατί ήρθε η ώρα να προβληματιστούμε σε σχέση με το τι γίνεται με το εμπόριο, τι γίνεται με τι επενδύσει και πώ μπορούν αυτέ τι δραστηριότητε να βελτιώσουν την κατάσταση με αυτέ τι αλυσίδε αξία, να βοηθήσουν σε κάποια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη για τους ε, οικονομικούς μας εταίρους και για την Ευρώπη βέβαια. Αυτές οι αλυσίδε, όπω είπατε έχουν καταστεί ένα κλειδί, ένα παράγοντα πολύ σημαντικό για την παγκόσμια οικονομία, ιδίω όσον αφορά την εμπορία και τι επενδύσει. Η διεθνή παραγωγή έχει ε, περισταθεί γύρω από αυτές τις ε, αλυσίδε και εκεί πέρα δρούν ε, με κάποιο είδους ε, δίκτυα οι πολυεθνικές, υπάρχουν ε, οι πάροχοι, οι θηγατρικές, οι εταίροι και κάποιοι μεμονωμένοι εργαζόμενοι και πάρα πολλές φορές δουλεύουν στον άτυπο τομέα και επίσης υπάρχουν και διαδοχικές υπεργολαβίες. Μιλούμε σήμερα για το 25% του παγκοσμίου εμπορίου και όπως είπατε το 75% του εμπορίου είχε να κάνει με αυτές τις αλυσίδε. Οπότε η νέα στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για επενδύσεις και εμπόριο, το εμπόριο για όλους αφορά αυτές τις αλυσίδε, επί τη βάση κάποιας ισόρροπης αντιμετώπιση για την επίτευξη των στόχων, δηλαδή το να ενισχυθεί η θέση της Ένωση στη διεθνή σκηνή, ε, σχέση με τρίτες χώρες, η βοήθεια για κινητικότητα, για υπηρεσίες και για το ψηφιακό εμπόριο, η πρόσβαση σε πρώτε ύλε, η προστασία τη καινοτομία και η αποτελεσματικότητα των τελωνιακών διαδικασιών. Αλλά αυτή η στρατηγική επίση θα πρέπει να πλαισιώνεται από περισσότερη υπευθυνότητα. Και για αυτό ο στόχο είναι να υπάρχει περισσότερη υπευθυνότητα από όλου του εμπλεκόμενου σε αυτέ τι αλυσίδε συμπεριλαμβανομένων ε, και των, των προσπαθειών για επιθετική πολιτική, για φορολογική πολιτική, για τις ε, προμήθειες και επίσης να υπάρχει κάποιο είδους ε, κοινωνική υπευθυνότητα αλλά και περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Το Κοινοβούλιο έχει συνθεί με την Επιτροπή σχετικά με αυτό και είπαμε ότι θα πρέπει το κεφάλαιο όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη να είναι εκταλεστό και σε σχέση με τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου, ελευθέρων συναλλαγών και να έχουμε μια διτή προσέγγιση. Να προστατεύσουμε το κοινωνικό πρότυπο αλλά και το κοινωτικό δίκαιο και από την άλλη μεριά να εξασφαλίσουμε βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση στην Ένωση και σε τρίτες χώρες. Καλούμε επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δείξει κάποιο είδου δεσμευτική δέουσα επιμέλεια και να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά αυτές τις αλυσίδες. Έχουμε αυτή την πρόσφατη, τον πρόσφατο κανονισμό ε, για τις συγκρούσεις και είπαμε ότι θα πρέπει να είναι η προσέγγιση δεσμευτικού χαρακτήρα. Οπότε η προσπάθεια μας αυτή εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Εκεί όπου η εμπορική πολιτική ε, ελκύει πολλέ επικρίσει από παντού. Και οπότε και γι' αυτό υπάρχουν πάρα πολλοί αυτοί που ε, θέλουν να αναδιπλωθούν. Και αυτό μας απασχολεί, αλλά ε, από την άλλη μεριά έχουμε και εκείνου οι οποίοι είναι θεμητό να θέλουν μια παγκοσμιοποίηση πιο δίκαιη, πιο διαφανή και Επίσης να έχουμε στο μυαλό μας την ε, Τζέντα 2030 και την ανάπτυξη για όλους. Οπότε ήρθε η ώρα να υπάρχει υπευθυνότητα, διαφάνεια και κοινωνική δικαιοσύνη όσον αφορά το περιβάλλον, όσον αφορά τα φορολογικά και έτσι να αποδείξουμε στους συμπολίτες μας ότι μπορούμε το εμπόριό μας να μας οδηγήσει ε, σε μια πιο δική Ευρώπη. Οπότε θέλουμε να έχουμε ένα τέτοιο ρόλο για τι παγκόσμιε αλυσίδε αξία και έχουμε ένα σωρό πρωτοβουλίε για διαφάνεια και για υπευθυνότητα. Έχουμε το βιώσιμο σύμφωνο για τον Παγκλαντέ, έχουμε τον κανονισμό για ορυκτά αιτία σειράξεων, ε, κανονισμό για τι πολυεθνικέ, αλλά επίση έχουμε τι κατευθυντήριε του ΟΗΕ. Ε, επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανάπτυξη των υποδομών και των τηλεπικοινωνιών, τη μείωση του κόστους εμπορίου και επενδύσεων λόγω των ε, πολιτικών ε, ε, απορρίθμισης και ε, επίση πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι γίνεται σε αναδυόμενε οικονομίε, Κίνα και Ινδία κυρίω. Δεν υπάρχει ομοιογενή ανάπτυξη αυτών των αλυσίδων σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν μεγάλε διαφορέ μεταξύ βιομηχανικών χωρών και των πιο φτωχών χωρών. Οπότε έχουμε τώρα κάποιες, κάποια προβλήματα, κάποιε προκλήσει για το περιβάλλον και όχι μόνο. Και ε, θα πρέπει να δούμε το ότι 50% των εμπορίων περνούν μέσω κάποιων ενδιαμέσων ε, σε κάποια, στην εμπορία τέλο πάντων στη δραστηριότητα μιας πολυεθνική, Οπότε οι βασικές ε, προκλήσεις για αυτές τις ε, αλυσίδε αφορούν τα κράτη, οι εμπορικέ πολιτικές, αυτές τις εταιρείε, οπότε έχουμε και προκλήσεις αλλά και ευκαιρίε για το εμπόριο και τις επενδύσεις, μείωση των δασμών, κανόνες προέλευσης, μορικές διευκολύνσεις, διαφάνεια, θεμητή δέος επιμέλεια, αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη όσον αφορά τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, εγκατακλείδη. Με αυτό το κείμενο έχουμε κάποιες συστάσεις για την εμπορική πολιτική και για τις επενδύσεις και έτσι να μπορέσουμε να έχουμε εμπόριο βιώσιμο και πιο δίκαιο να υπάρχουν κάποιες προβλέψεις ε, σε συμφωνίες συναλλαγών δεσμευτικέ, να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή των πολυεθνικών, γιατί για να αποφύγουν φόρου χρησιμοποιούν ακριβώ αυτέ τι ε, αλυσίδε. Ε, να δούμε τι γίνεται με αυτά τα ορυκτά σειράξεων ε, και να προτείνουμε κάποιες ε, πρωτοβουλίες για την δέουσα επιμέλεια όσο πρέπει την αλυσίδα προμήθειας των πολυεθνικών. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Δίνω το λόγο στους κύριους συζητητές για το ΕΛΚ. Κύριος Βαλέντσα, του κύριου Μπάλσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο συνάδελφος Φερνάντο είχε κάποια πολιτικού χαρακτήρα που χρήσε στην Πορτογαλία και δεν μπορούσε να προσέλθει, αλλά ε, προτίμασε μια ομιλία την οποία θα ήθελα να σα διαβάσω, αν μου επιτρέπετε. Ε, καταρχήν ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω, μα αναφέρει για ο συνάδελφος, τη συνάδελφο για αυτό το έγγραφο εργασία που μα υπέβαλε και το οποίο μπορεί να αποτελέσει μια καλή βάση για τι εργασίε που θα ξεκινήσουμε σήμερα σε ό,τι αφορά την έκθεση με την γνωμοδότηση πρωτοβουλία που θα ακολουθήσει. το ζήτημα των παγκοσμίων λοιπόν αλυσίδων αξία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε διαφορετικά επίπεδα και με διαφορετικά μέσα. Για παράδειγμα, θα πρέπει να δούμε ε, να δούμε το τι συμβαίνει ε, ε, σε ό,τι αφορά το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικά τη παγκόσμια οικονομία και το πώ διαμορφώνονται αυτέ οι αλυσίδε παγκοσμίω. Ε, τα ζητήματα της, ε, του σεβασμού του περιβάλλοντο, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, αλλά και οι ανάγκε τη περαιτέρω ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασία αποτελούν τμήματα μια γενικότερη στρατηγική βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, Τη προστιμένη αξία ε, μέσω των ε, επιχειρήσεων, ειδικότερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και η λήψη υπόψη του ταχαίως μεταβαλλόμενου συστήματος διαχείρισης των επιχειρήσεων ε, που έχουμε σημαίνει ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με συνεχώς ε, διαφορετικές ε, πραγματικότητες. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν διαστάσεις τις οποίες θα πρέπει πάντοτε να έχει κατά νου η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ώστε να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που συνοδεύουν αυτές τις αυτή την πραγματικότητα. Και το κάνει ήδη, για παράδειγμα, μέσω ε, της ε, ε, κοινή πρωτοβουλία και με τον Μπαγκλαντές και με, τη, το Μιανμάρ, και με τη Μιανμάρ, αλλά και μέσω του κανονισμού, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την παράνομη νοοτομία και το κανονισμό για τα βιοκαύσιμα. πέραν αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε τα εξή. Θα πρέπει να γνωρίζουμε την περιπλοκότητα και την ταχαίως μεταβαλλόμενη το, το μεταβαλλόμενο χαρακτήρα των ε, παγκόσμιων ε, αριστερών αξία. Δηλαδή τα συστήματα παραγωγής τη σήμερα ημέρα είναι εξαιρετικά περίπλοκα και ε, περιλαμβάνουν μία σειρά από διαφορετικά δίκτυα τα οποία μεταβάλλονται σε ό,τι αφορά τα επιχειρηματικά τους μοντέλα. Αυτό επιτρέπει την ταχαία, διασυνοριακή εμπορική ανάπτυξη. Οι κινητήρες δυνάμει είναι διαφορετικές δηλαδή οι δυνάμεις αυτών των αλυσίδων αξίας, αλλά κάποιες από αυτές είναι μετρήσιμες και κάποιες όχι, όπως αναφέρεται και στη σχετική μελέτη της ε, Παγκόσμιας Τράπεζας. Και η Επιτροπή ε, στην ε, εμπορική της στρατηγική εμπορού για όλους αναφέρει ότι θα πρέπει να να ε, συμπεριλάβουμε ε, ε, στην διαμόρφωση αυτή τη στρατηγικής σε μία σειρά από φορεί σε περιφερειακό, τοπικό και εθνικό και ενωσιακό επίπεδο και θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας το πόσο ε, γρήγορα μεταβάλλονται οι σχετικές ε, αλυσίδες αξίας με βάση τα όσα συμβαίνουν για παράδειγμα πρόσφατα με τις ε, εκλογές στην ΕΠΑ, με την απόφαση για το Brexit και την ανάδυση νέων οικονομικών φορείων αλλά και την αστάθεια στην Μέση Ανατολή, τις ανισότητες που υπάρχουν, τις μεταναστευτικές δροές, τις τρομοκρατικές απειλές, τα αέρα του θερμοκηπίου, την περιβαλλοντική υποβάθμιση αναβάθμιση, ε, την επιβολή του σύγχρονου τρόπου ζωής, του ε, τους καινοτόμους ε, διάβλους ροής πληροφοριών. Όλα λοιπόν αυτά τα στοιχεία αυξάνουν ακόμα περισσότερο την περιπλοκότητα της σημερινής πραγματικότητας. Πέραν αυτού θα θέλαμε να γίνουν πιο συγκεκριμένες αναφορές σε ό,τι αφορά τον κέριο, την κέρια σημασία των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις ε, παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Θα πρέπει ε, να αναφέρουμε την ανάγκη για την προώθηση ποιοτικών ε, θέσεων εργασία και την ανάγκη του να μην εγκαταλείπουν του χώρου στου οποίου διαβιούν οι πολίτε. Επίση, θα πρέπει να υπάρξουν πολιτικέ οι οποίε θα υποστηρίξουν αυτέ τι μικρομεσαίε επιχειρήσει να συμβάλλουν σε αυτέ τι ε, παγκόσμιε αλυσίδε αξία, ειδικότερα στι χώρε εκείνε με χαμηλό εισόδημα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν αυτέ οι επιχειρήσει θα μπορέσουν να συμμετάσχουν περισσότερο στι παγκόσμιε αλυσίδε αξίε που εκπροσωπούν σήμερα το 75% του παγκόσμιου εμπορίου. Επίση, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε το πόσο σημαντικό είναι να ε, ε, εξαλείψουμε τα context costs όπως αναφέρονται δηλαδή ε, ε, κάποιες δαπάνες οι οποίες λειτουργούν αποτρεπτικά σε ό,τι αφορά ακριβώς αυτή τις, ε, την εμπλοκή της ενεργό συμμετοχής της ε, ε, αλυσίδας αξίας. Και εδώ αναφερόμαστε ειδικότερα σε ζητήματα επιμελητίας, στην έλλειψη προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ανεπαρκής ρήτρες σε ό,τι αφορά τις θέσεις εργασίας και ούτω καθεξής. Από εκεί και μετά καλούμε να υπάρξει καλύτερη εφαρμογή των σχετικών ε, προτύπων σε ό,τι αφορά την εταιρική ευθύνη και τι ε, θέσει εργασία ε, που έχουν προωθεί από, τις, από του σχετικού παγκόσμιου οργανισμού. Θα ήθελα σε αυτό το πλαίσιο να υπογραμμίσω και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μαΐου του 2016, όπου υπογραμμίζεται η σημασία της εφαρμογής αυτών των μέτρων, καθώς προωθεί την βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημιουργία σταθερών μονίμων θέσεων εργασία και περισσότερη, περισσότερο empowerment για όλους ειδικότερα για τους νέους ε, και για τις γυναίκες αλλά και για ε, ευάλωτες ομάδες όπως άτομα με αναπηρία. Με την υποστήριξη λοιπόν ε, της εφαρμογής ΕΣΑΤ θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ε, κάποιες ε, προτάσεις που είχαμε συμφωνήσει πέρσι τον Ιούλιο σε ό,τι αφορά δηλαδή το ψήφισμα σε ό,τι αφορά το εμπόριο και τις επενδύσεις ε, και τις, το ψήφισμα σε ό,τι αφορά τις συστάσει του 2010 σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ευθύνη των επιχειρήσεων. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να τονίσω το πόσο σημαντικό είναι στις μελλοντικέ εμπορικέ συμφωνίε να λαμβάνονται πάντοτε υπόψη περιβαλλοντικά ζητήματα και ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και δεσμεύσεις σε ό,τι αφορά ε, δικαιώματα εργασίας, όπως αυτά ε, εκπηγάζουν και από τις ε, συμφωνίε σε επίπεδο Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας. Και υπενθυμίζω την το δικό μας κάλεσμα προς την ε, Επιτροπή να συνεχίσει τις ε, προσπάθειές της για περισσότερη ανάληψη ευθύνης από την πλευρά των επιχειρήσεων, ε, οι οποίες θα πρέπει να σέβονται πλήρως τις, τα πρότυπα της ΆΕΛΟ αλλά και τα πρότυπα CSI ειδικότερα. Όμως αυτά έχουν διατυπωθεί από τον ΟΣΑ, τα Ηνωμένα Έθνη, και τις κατευθυντήρες γραμμές ΑΕΣΟ και ΑΕΛΟ ειδικότερα στους, ε, στο, στο υφαντουργίας ε, και της εξωτερικής βιομηχανίας. Ε, κλείνοντας, να πούμε ότι θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες ε, προκειμένου να υπάρξουν πιο σαφείς αναφορές πιο αναφορές σε ό,τι αφορά την προώθηση πολιτικών ε, για την καταπολέμηση της καταναγκαστικής εργασίας και της εμπορία ανθρώπων που δεν αναφέρεται πουθενά ρητά στο κείμενο και επίσης ε, θα θέλαμε να υπάρξει, να αναφερθεί περισσότερο μια ολιστική προσέγγιση σε ό,τι αφορά το φύλλο, το οποίο ως ζήτημα το φύλλο αναφέρεται μόνο σε τέσσερις σειρέ Αυτό το εγγράφου. Επίσης θα κάνουμε λόγο για την ανάγκη ιδιαίτερης εστίαση σε ειδικέ ευάλωτες ε, ομάδες ατόμων όπως ε, επανέως άτομα με αναπηρία και βέβαια αναμένω ε, με ενδιαφέρον την ε, περαιτέρω εξέταση αυτών και άλλων ε, προκλήσεων από κοινού με τον εισηγητή και τους κοιόδες εισηγητής σε ό,τι αφορά το ζήτημα των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας, όπως για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τους κανόνες καταγωγής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και αναμένω με ενδιαφέρον και την πρόταση ψηφίσματος που ακολουθήσει. Yeah. Ο κύριος Λόνς δεν είναι εδώ. Θέλετε εσείς να μιλήσετε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος της ομάδας μου. Θα ήθελα να πω τα εξή. Βεβαίως ε, ζούμε σε έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης και έχουμε παγκόσμια αλυσίδα αξίας. Ε, προϊόντα σχεδιάζονται σε μία χώρα, κατασκευάζονται σε άλλες, ε, συναρμολογούνται σε παράλλες και υπάρχουν διάφορα επίπεδα ανισορροπιών που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Εμείς ως ομάδα είμαστε υπέρ ε, της εισαγωγής ε, πρακτικών που θα μας βοηθήσουν να καταπολεμήσουμε ε, τέτοιες χρηματοπιστωτικές ροές για να καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή, ε, που βοηθούν άλλες ε, παράνομες πρακτικές, να υπάρχει διαφάνεια. Έχουμε όμως ε, πολλές δυνατότητες για να εισαγάγουμε δεσμευτικά κεφάλαια βιώσιμης ανάπτυξη, κυρώσεων, στις προτάσεις για εταιρική κοινωνική ευθύνη. Πότε; δεν ήμασταν υπέρ μιας στρατηγικής ε, όρων ή προπετούμενων ή κυρώσεων. Εμείς ε, προωθήσαμε και προτιμούσαμε μια στρατηγική εμπλοκής όπου θα αντιμετωπίζουμε τους ε, εμπορικούς μας εταίρους επίσης όρους. Και όταν μιλάμε για κοινωνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές, θεωρούμε ότι και οι χώρες χρειάζονται τέτοιες προδιαγραφές που θα ανταποκρίνονται στο δικό τους επίπεδο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και οποιαδήποτε προσπάθεια να επιβάλλουμε τις ε, δικές μας ε, τις προδιαγραφές θα είναι αντιπαραγωγικές και τελικά θα σημαίνουν ε, άλλη μια μορφή προστατευτισμού. Επίσης, όταν μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα, εργατικά δικαιώματα και όλα αυτά τα σημαντικά θέματα Έχω την αίσθηση ότι η ίντα πραγματικά θα πρέπει να είναι μια πλατφόρμα συζήτησης για άλλες πτυχές ε, του εμπορίου και έχουμε νομίζω εδώ άλλες επιτροπές στο Κοινοβούλιο που θα συζητηθούν αυτά τα ζητήματα. Δυστυχώς αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ στην Επιτροπή μας συχνά είναι αντίθετο με αυτό το οποίο θεωρούμε ότι θα πρέπει να συμβολίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τη διεθνή συνεργασία και το ελεύθερο εμπόριο. Και το να θέτουμε σε εμπόδια ή προαπαιτούμενα δεν είναι σωστό. Δεν πρέπει να αναζητούμε προφάσεις για προστατευτισμό. Τέλος, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι παγκόσμιες αυτές αλυσίδες αξίες έχουν κάποιον αντίκτυπο στην οικονομία. Αφενό για τις αναψώμενες χώρες ε, το να ανταχθούν σε μια τέτοια αλυσίδα σημαίνει ξένε επενδύσεις και άρα έτσι, οι δασμοί άλλα τέτοια εμπόδια γίνονται περιτά γιατί η φορολόγηση εισαγόμενων εξαρτημάτων, απλά ξανά το κόστος. Θα πρέπει λοιπόν ε, να σκεφτούμε να μειώσουμε αυτά τα, αυτούς τους φραγμούς στο εμπόριο όπως ε, τους δασμούς ε, κτλ. Από την άλλη έχουμε αναπτυσσόμενες χώρες που πρέπει επίσης να προσαρμοστούν γιατί πολλές αμφισόμενες χώρες ε, πήγαινουν στην κατεύθυνση της υποκατάστασης ε, εισαγωγών. Όλοι ξέρουν πως βεβαίω ο η παραδοσιακή βιομηχανία είναι πολύ σημαντική, αλλά οι θέσει εργασία ε, δεν θα επιστρέψουν σε αυτές τις βιομηχανίες, οι οποίες είναι πολύ κερδοφόρες, αλλά λιγότερο από το παρελθόν. Και άρα πρέπει να εστιάσουμε και στις υπηρεσίες που σχετίζονται με την παραγωγή, σχεδιασμό, λογισμικό κτλ. που οπωσδήποτε θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Θα παρότεινα λοιπόν να δούμε και αυτά τα ζητήματα λεπτομερώς στην έκθεση αυτή. Αυτά. Για την ώρα αναμένουμε τις περαιτέρω συζητήσεις και είμαστε στην διάθεσή σας για συνεργαστούμε. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Ζάχραντιλ, για την Άλτε, η κυρία Σάραντσεβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θεωρώ θετική αυτή την εκθεσία της πρωτοβουλίας, να ευχαριστήσουμε και την εισηγήτρια για τη δουλειά τη γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι αλυσίδες αξίας για την οικονομία, για το εμπόριο, άρα και θα πρέπει να υπάρχει κάποιο είδου ολοκληρωμένη προσέγγιση. Ακριβώ αυτό το οποίο υποστηρίζει ε, στο έγγραφο η συγγήτρια που τονίζονται ε, όλες οι πλευρές, ε, το πώς θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, το πώς θα πρέπει να είναι σεβαστές οι ενωσιακές αξίες, οπότε ακριβώς αυτά είναι τα θέματα που αντιμετωπίζουμε σε σχέση με το εμπόριο. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για κάθε στρατηγική σχέση με το εμπόριο. Αυτό θα πρέπει να καλύψει όλου του τομεί του εμπόριου και τι ε, αλυσίδε αξία. Άρα θα πρέπει να εστιάσουμε τώρα στο πώ θα είμαστε πιο δυναμικοί, πιο δραστήριοι, ούτω ώστε να δοθούν ευκαιρίε μέσω ε, αυτή τη ρύθμιση και ε, για το εμπόριο και για του εργαζόμενου. να μην είμαστε απλώς τιμωρητικοί, ε, αντί για αυτό που λέει για τα δεσμευτικά μέτρα, να δούμε πώ μπορούμε να εκμεταλλευτούμε πλήρω τι προσφερόμενε ευκαιρίε που προσφέρονται με τι αλυσίδε αξία. Η κατάτμιση στην παραγωγή έχει δημιουργήσει πολλέ ευκαιρίε Φερρυπίν για τι ε, ΜΜΕ στην Ευρώπη, από πλευρά των τέρνων για να έχουμε πρόσβαση σε διάφορε αγορέ για τις αλυσίδες ε, αξίες. Άρα αυτό να ερευνήσουμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα περιβάλλον όπου να μπορούν οι ΜΜΕ να συμμετάσχουν σε αυτές τις ε, αλυσίδες. Πώς μπορούν να ενταχθούν στις παγκόσμιες αγορές. Εδώ το έγγραφο θίγει διάφορα σημαντικά ζητήματα για τις αλυσίδες αξίες, Φερρυπίν το πώς θα πρέπει ταχείας οι ικανού διευκόλυνση του ΠΟΕ να υλοποιηθούν. Υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία όμω τα οποία φαίνονται προβληματικά. Φερρυπίν, εκεί που λέει ότι η έλλειψη διαφάνεια ε, όσον αφορά τι αλυσίδε ε, οδηγούν σε ε, καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προτύπων. Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο να το αναφέρουμε εδώ, όσον αφορά τη συμμετοχή στι αλυσίδε, γιατί τα υπέρνει πολύ πολύ περισσότερα από τα κατά τέλο πάντων από τέτοιου φόβου, όπω εδώ αυτέ οι αλυσίδε ε, είναι πηγή απασχόληση ε, εισοδήματο σε πολλές αναπτυσσόμενε χώρες και έχουν βγάλει από τη φτώχεια εκατομμύρια. Άρα θα πρέπει να δούμε τώρα πώς θα συνεχίσουμε το να μπορούμε να μοιραστούμε τις ε, καλύτερε αρχές και αξίες με τους εταίρους μας, να υπάρξουν κίνητρα με το σύστημα εγγεμένων προτιμήσεων πλάς, όπως είπε και η συγκέντρια, να δούμε πώς θα αναθεωρηθούν οι κανόνες προέλευσης, αλλά βέβαια το ισχυρό σύστημα λειτουργεί μια χαρά. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει και πώς θα βοηθήσει τώρα έχουμε εδώ πέρα και κάποιους κανόνες για την ισότητα των φύλων. Είναι αλήθεια ότι θα πρέπει να μην υπάρχουν μυρωδής αναλογία για τα ωφέλη μεταξύ ανδρών και γυναικών από αυτά, και να υπάρξει ρύθμιση ανά κλάδο, ανά τομέα. Πολλές φορές ε, οι γυναίκες ε, ε, αδικούνται δύο σαν τις χώρες. Αλλά με την εμπορική πολιτική δίνονται αυτά τα προβλήματα. Δεν έχουμε αρκετά στοιχεία όσον αφορά το πώς η εμπορική πολιτική και το εμπόριο επιδρούν στην ισότητα των φυλών. Άρα θα πρέπει να ξεκαθαριστούν αυτές οι προτάσεις. Επίσης η επέκταση των ε, κανονισμών για τη δοσητική οργανισμού Βρυξέλλες ε, παρθμόν 1 ε, και αυτό είναι σημαντικό θέμα που θίγεται οπότε και ευχαριστώ πάρε την συγκίτρια και προσλέπω στην συνεργασία την Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να ευχαριστήσω την συγκίτρια διάβασα με μεγάλο ενδιαφέρον το έγγραφο Είμαι ικανοποιημένη με την προσέγγιση που έχει αυτή η έκθεση για τις θετικές και αρνητικές πτυχές του διεθνούς εμπορίου. Και συμφωνώ με τις αφετηρίες της. Ε, θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια δεσμευτική πρωτοβουλία για το due diligence και επίσης ε, δεσμευτικές ρήτρες για την βιώσιμη ανάπτυξη. Και πρέπει να πω ότι με εξέπληξε θετικά και η στάση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Αλλά αυτό το οποίο δεν βλέπω εδώ είναι μια θεμελιώδης ανάλυση των τεράστιων διαφορών που υπάρχουν μεταξύ φτωχών και πλούσιων χωρών. Στον κόσμο βεβαίω καλό και αναγκαίο είναι να δούμε τι γίνεται με την επιμέλεια την διαφάνεια, τη διάσταση του φίλου, αλλά εάν δεν πάμε πιο βαθιά από αυτό θα μεγαλώσουν μόνο οι διαφορές. Όταν υπάρχει. Ε, οργανώνουμε έναν αγώνα μεταξύ ποντικών ε, και ελεφάντων. Πρέπει να προστατεύσουμε βέβαια, αλλά δεν αρκεί να λέμε ότι θα προστατεύσουμε τα ποντίκια. Πρέπει να αποφύγουν πρώτα απ' όλα τα ποντίκια το να μην τα πατήσουν οι ελέφαντες. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τα θέματα του περιβάλλοντος, του κλίματος, ε, πράγματα τα οποία προκαλούν πείνα και δυστυχία και στέλνουν μετά πρόσφυγες στις δικές μας χώρες. Πράγματα τα οποία βλέπουμε και μετά από τη δικιά μας την πλευρά εξυπνούν καταστάσεις λαϊκιστικές και εθνικιστικές. Θα πρέπει λοιπόν να καταλήξουμε σε έναν περιορισμό του παγκοσμίου εμπορίου και θα πρέπει Βεβαίω να πούμε ότι για αυτούς οι οποίοι λένε ότι οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές διατάξεις είναι μέτρα περιοριστικά του εμπορίου, αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να βάλουμε δασμούς στα προϊόντα εκείνα τα οποία δεν πληρούν περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς όρους και τα λεφτά αυτά να πηγαίνουν σε ένα ταμείο για να βοηθήσουν τις χώρες αυτές να εκπληρώσουν αυτές τις χώρες. Να μην τις τιμωρούμε δηλαδή, αλλά να επενδύσουμε, να έχουμε μια διαρθρωτική λύση. Νομίζω είναι το απλούστερο μέσο που έχουμε για να μπορέσουμε να κατευθύνουμε κάπως το παγκόσμιο εμπόριο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. το λέγεται Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τη Μαρία Αρένα για το ενδιαφέρον αυτό εγγραφό εργασία και νομίζω ότι είναι μια χρήσιμη αφετηρία η στρατηγική εμπόριο για όλους, η οποία αναφέρει συγκεκριμένα τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας ε, και το πώς θα πρέπει να προωθήσουμε έτσι την παγκόσμια διακυβέρνηση και δεν βλέπω πώς αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε το εμπόριο είναι απλά εμπόριο και δεν έχει ουδεμία σχέση με την ανάπτυξη ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Και Θεωρώ ότι η αναφορά στην Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ μας δείχνει ότι πρέπει να ενσωματώσουμε διάφορους τομείς ε, πολιτικής για να απαντήσουμε στις παγκόσμιες προκλήσεις. Αλλά προφανώς, όπως ε, λέει ο συγητής, οι αλυσίες αυτές ε, δεν ωφελούν εξίσου τους διάφορους δρόντες ε, και φορείς. Γι' αυτό ακριβώς ε, θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα για να συμμετέχουν και αναψώμενες χώρες ε, και επιχειρήσεις τους και δεν μπορώ να σκεφτώ εγώ κάποιο καλύτερο θεσμικό όργανο από το Διεθνές Κεντροπορείο του ΠΟΕ που επί σειρά ετών προωθεί το ε, Aid for Trade. Θεωρώ λοιπόν πως έχει φτάσει η στιγμή να δούμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ακολουθήσει μια ολιστική πρωτοβουλία για υποχρεωτική μέλη όπως προτείνει η κυρία Αρένα. Έχουμε διαφορετικές ε, τομεακές ε, πρωτοβουλίες και όπως σημειώνει κάποια κράτη-μέλη έχουν ήδη επιβάλλει τέτοια νομοθεσία όπως ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γαλλία και δεν είναι η μόνη και θεωρώ ότι λόγω της ε, πίεσης του κοινού για να δούμε το, πλαίσιο σε ένα, το εμπόριο σε ένα συνολικότερο πλαίσιο θα δουν περισσότερα τέτοια εκτός αν κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Κομισιόν τι συνέβη με την πρωτοβουλία για την ανακοίνωση της Κομισιόν για το σχέδιο δράσης για την υπεύθυνη συμπεριφορά των επιχειρήσεων, το οποίο περιμένουμε εδώ και 1,5 χρόνο, γιατί έχει κολλήσει στην Κομισιόν. Περιφέρεται μεταξύ διαφόρων γενικών διευθύνσεων που δεν μπορούν να συμφωνήσουν. Οι προτάσεις λοιπόν στο έγγραφο αυτό πραγματικά αξίζει να εξεταστούν καλύτερα και στενότερα και είναι ενδιαφέρον ότι ο συγητής προτείνει να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογή της οδηγία Βρυξέλλες 1 για τους κανόνες δικαιοδοσίας για να ισχύουν για τρίτες χώρες σε περιπτώσεις ε, κατά εταιριών που έχουν ε, την έδρα τους ή σημαντικό μέρος το, το, της δραστηριότητάς τους εκτός της Ένωσης. Πρέπει να το δούμε λοιπόν. Και βεβαίως ε, έχουμε το πολύ ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα του πώς ε, θα μπορέσουμε το εμπόριο να είναι υποφελές για όλους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω την ε, Μαρία Ρενά γιατί και αυτή τη φορά το κείμενό της είναι άριστο. Το διάβασα δε με μεγάλο ενδιαφέρον και σχεδόν 100% σύμφωνο σήμερα. Στηρίζεται το εμπόριο σε αυτές τις αλυσίδες αξίες που ξαπλώνται σε ολόκληρες πύρους. Ένα κινητό δεν είναι απλώς κινέζικο. Έχει από όλο τον κόσμο διάφορα ε, κομμάτια και όμως πολλές φορές δεν ωφελούνται όλοι ε, αυτές οι αλυσίδε. Είναι αλήθεια στις τελευταίες δεκαετίες είχαμε ανάπτυξη. Παγκοσμίω υπήρξε ένα, ε, ένα άνοιγμα ε, αλλά πολλές φορές μεγάλωσαν και οι ανισότητες και αυτό το οποίο χρειάζεται να καταλάβουμε ότι θα πρέπει το εμπόριο να γίνει όργανο όχι μόνο ανάπτυξη, αλλά και εργαλείο ε, της τη περιθωριοποίηση, τη κοινωνική. Ε, Επομένω, θα πρέπει πέραν των οικονομικών να δούμε και τι θα γίνει από πλευρά ανθρώπου και ε, έτσι θα ε, ωφελήσει αυτή με πάρα πολλέ χώρε πόλη ανάπτυξη, έχουν τέτοιες αλυσίδες αξίας οι οποίες θα πρέπει ακριβώς τέτοια ανάπτυξη βιώσιμη να ε, προωθούν και να μην είναι απλώς χώρος με την κατάσταση από τις πλούσιες χώρες. Άρα θα πρέπει να έχουμε εδώ πέρα ε, για την βιώσιμη ανάπτυξη κάποιες ε, συστάσεις δεσμευτικές και όχι μόνο δηλώσεις αρχής. Κάποιε κυρώσει για αυτού που δεν σέβονται την εργατική νομοθεσία αλλά και την περιβαλλοντική νομοθεσία. Συμφωνώ επίση και όταν λέμε για κάποιο είδου ανεξάρτητε ελεγκτικέ αρχές που επιβάλλουν αυτέ τι ε, κυρώσει, όταν υπάρχουν ε, καταχρήσει, παραβάσει και για την επιχείρηση αλλά θα πρέπει να ε, τηρούνται και διάφορες ρήτρε όσον αφορά τις χώρες με τις οποίες έχουμε εμπορικές συμφωνίες. Ε, Επομένω να ελέγχεται ότι γίνεται από ανθρωπίνων δικαιωμάτων και Περιφάλλοντο. Σωστή αυτή η έκθεση πρωτοβουλία και πιστεύω ότι η συγκίτρια θα προωθήσει εδώ, θα έχουμε τέτοια στρατηγική, θα φτάσει η έκθεση στην Ολομέλεια. Και επίσης έχουμε και αύριο να εγκρίνουμε κάποια έκθεση όσον την τελειωνική νομοθεσία και ελπίζω ότι έτσι θα υλοποιήσουμε αυτά τα οποία έχουμε εξαγγείλει. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλησπέρα. Τέθηκαν μια σειρά από ερωτήματα προς την Επιτροπή. Οπότε καταρχήν επιτρέψτε μου από την πλευρά μας να ευχαριστήσουμε τον είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και αυτή την νομοδότηση. Έχουμε συναδέλφους εδώ από τη φίσμα την Growth, εγώ είμαι από την Trade, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα για εμάς και αναφερθήκατε ε, σε μία σειρά από θέματα τα οποία δεν καλύπτονται μόνο από το θεματολόγιο, το εμπορικά θεματολόγιο, αλλά καλύπτουν και μία σειρά από περαιτέρω ζητήματα. Πράγματι, τα όσα αναφέρετε καταδεικνύουν το εύρος και το βάθος της εν λόγω συζήτησης, δηλαδή οι διάφοροι δίευλοι οι οποίοι εμπλέκονται στις ε, αλυσίδες αυτές της αξίας και το πώς και εμείς θα πρέπει να προσαρμόσουμε ανάλογα τις δικές μας πολιτικές. Ήδη ε, κάνουμε πολλά και να αναφερθώ σε κάτι για το οποίο είναι αρμόδιος ο συνάδελφος εκτεξιών ε, δηλαδή ε, αυτός ο κανονισμός σε ό,τι αφορά το non-financial disclosure, δηλαδή ε, την διάθεση πληροφοριών από την πλευρά μεγάλων ομίλων σε ό,τι αφορά πολιτικές σε σχέση με περιβαλλοντικά ζητήματα, δικαιωμάτων ε, των εργαζομένων, ε, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταπολέμηση της τοροδοκίας. Η πρώτη έκθεση ε, προβλέπεται μάλιστα να υποβληθεί το 2018. Ο συνάδελφος μπορεί να σας δώσει και περαιτέρω πληροφορίες. Από εκεί και μετά έχουμε και πιο πρόσφατη νομοθεσία σε ό,τι αφορά νέες διατάξεις, σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις για την ε, καλύτερη ακριβώ ε, συμμόρφωση με τις σχετικές ε, προϋποθέσεις. Από εκεί και μετά και η Γενική Διεύθυνση αλλά και η ΔΕΦΚΟ έχουν ξεκινήσει σε ό,τι αφορά το capacity building αλλά και τη δημιουργία περαιτέρω προγραμμάτων και από εκεί και μετά και, άλλες, και η εξωτερική υπηρεσία και άλλες γενικές διευθύνσεις έχουν ξεκινήσει δράσεις συνεργασίας με τρίτες χώρες παραγωγής και προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε τα όσα έχουμε στο κεκτημένο, για παράδειγμα ε, μέσω του συστήματος ε, γενικεμένων προτιμήσεων Plus, ε, να δημιουργήσουμε περαιτέρω όθηση αυτέ τι αξίε βασιζόμενη και στα όσα έχει κάνει και εδώ και ο, και Παγκόσμια Οργάνωση Εργασία, ε, τα όσα έχουν επιτευχθεί στο πλαίσιο συμφωνία με τον Παγκλαντέ και ό,τι καθεξή. Και εμεί ε, προφανώ ε, θέλουμε να προωθήσουμε περισσότερο την ε, πτυχή τη βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο των εμπορικών μα συμφωσιών, δηλαδή θέλουμε να δώσουμε και περισσότερη έμφαση στη δέσμευση ό,τι αφορά την ανάληψη ευθύνη από πλευρά των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, έχουμε ξεκινήσει και ένα χώρο που ε, την και τον, τον ΩΣΑ ακριβώς για το ζήτημα της ε, ε, ε Επίση, Επίσης ε, προσπαθούμε να δούμε πώς ε, μπορούμε να εφαρμόσουμε καλύτερα τα κεφάλαια TST στο πλαίσιο των συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου. από εκεί και μετά, ποιες είναι κύριες αρχές που διέπουν τις δικές μας εργασίες. Καταρχήν θέλουμε να έχουμε ένα έξυπνο συνδυασμό πολιτικών. Συμφωνώ δηλαδή με μια σειρά από ομιλητέ ε, που είπαν ότι είναι ταχαίω μεταβαλλόμενος ε, αυτό ο τομέα. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, το κατάλληλο e ευφυέ συνδυασμό πολιτικών. Επίση θα πρέπει να οικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ των συναρμόδιων φορέων και να δούμε και να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι ο καθένας είναι ο πλέον ενδεδειγμένος για να γνωρίζει το πώ θα εφαρμόσει τι ειδικές άρχες. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε τις συμμαχίες με τους ε, ε, σχετικούς ε, εταίρους που έχουμε και στις τρίτες χώρες και με τις σχετικές επιχειρήσεις. Γιατί χωρίς να υπάρξει τέτοια καλύτερη συνεργασία και περισσότερη εμπιστοσύνη δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις σχετικές πολιτικές. Δεν είμαστε δηλαδή εμείς ο μόνος εμπορικός εταίρος των τρίτων χωρών. Υπάρχουν και άλλοι. Δεν θα πρέπει να σταματήσουμε την επαφή μας και τις συνεργασίες μας με χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα ε, Πρόκειται δηλαδή για χώρες οι οποίες ακριβώς βασίζονται σε εμά και σε άλλους προκειμένου να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Οπότε χρειαζόμαστε λοιπόν ε, μια κουλτούρα αν θέλετε εδώ η οποία ε, δεν επιτρέπει αποκλεισμού. Και από εκεί και μετά μου επιτρέπετε θα δώσω το λόγο στον Εντουαρτούν από την Γενική Διεύθυνση Growth καθώς ε, τέθηκε και ένα συγκεκριμένο ερώτημα στο συνάδελφο. Και από εκεί και μετά και ο συνάδελφο από την Εφήσμα μπορεί να δώσει περαιτέρω διευκρινήσει σε ό,τι αφορά ε, τον κανονισμό για ε, τις σχετικέ πληροφορίε των non-financial disclosure. Ευχαριστώ και εγώ από την πλευρά μου και την εισηγήτρια και την κυρία Χάουταλα για τα ερωτήματα. και την όλη συζήτηση που έχει ξεκινήσει και στο επίπεδο της Επιτροπής και να πω ότι εμείς ε, στην Κομισιόν, στην Κομισιόν όχι μόνο στην DG η Κομισιόν έχει αποφασίσει σε αυτή τη φάση να δώσει περαιτέρω πολιτική όθηση στην εφαρμογή της ατζέντα των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που εγκρίθηκε πριν από ένα χρόνο στο ΟΗΕ το Νοέμβριο έκανε μια ανακοίνωση που περιλαμβάνει όλες τις πολιτικές, όλες τις πρωτοβουλίες ε, που θα συνεισφέρουν σε μια σειρά ζητημάτων αηφορίας. τις δράσεις αυτές ε, που αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε ήδη από το 2011. Δεν το έχει αναφέρει κάποιος άλλος. Ο ότι όλα αυτά τα μέτρα περιλαμβάνονται στην ε, στρατηγική εταιρική κοινωνική ευθύνη που εγκρίθηκε το 2011 και αναφέρονται σε όλες τις γραμμές του ΟΣΑ, του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας ε, και αυτή τη στιγμή εμείς ε, προσπαθούμε να εφαρμόσουμε αποτελεσματικά όλα τα μέτρα που υπάρχουν εκεί η οδηγία για τις δημόσιες προμήθειες, για τα δικαιώματα των μετόχων που συμφωνήθηκε στον τριμερή διάλογο, ο κανονισμός για τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων, μέτρα αποφυγής της φοροδιαφυγής, όλα αυτά τα οποία ακόμα συζητούνται σε διάφορες επιτροπές του Κοινοβουλίου οπότε υπάρχουν διάφορα νομοθετικά μέτρα που περιλαμβάνουν αυτά τα οποία είπαν οι συνάδελφοι δηλαδή τις ευέλθες πρακτικές ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τις υπεύθυνες επιχειρήσεις, πολλά βέβαια πράγματα λοιπόν, τα οποία θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε. Επίσης δεν αναφέρθηκε, η Κομισιόν ξεκίνησε μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία λέγεται βιώσιμη χρηματοδότηση μια ομάδα υψηλού επίπεδου με τους κύριους επενδυτές για να πείσουμε την επενδυτική κοινότητα να εμπλακεί πολύ περισσότερο στις αποφα... και να ενσωματώσει στις αποφάσεις τους, ε, να ενσωματώσουν κριτήρια κοινωνικά κτλ. Οπότε εμείς ε, υλοποιούμε όλες τις δράσεις που είχαμε ήδη καθορίσει το 2011. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο δράσης αυτή τη στιγμή δεν δεν είναι το μεγάλο θέμα γιατί το Νοέμβριο του 2016 στην ανακοίνωση είχαμε ανακοίνωση ότι η Κομισιόν θα εντείνει το έργο της και εξετάζουμε ιδιαίτερα γιατί εσείς ε, και η κυρία Ρένα το αναφέρατε το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε την επόμενη Τρίτη και θα έχουμε μια συγκεκριμένη εκδήλωση θα εντείνουμε ε, τη δουλειά μας παρακολουθούμε τη δουλειά μας ε, σε δύο κράτη-μέλη ε, η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία είναι οι δύο μόνες χώρες οι οποίες μέχρι στιγμής έχουν νομοθετικό κείμενο για το θέμα της δέουσας ευμέλειας. Θα παρακολουθούμε αυτά στενά ε, καθώς δεν έχουμε ακόμα ξεκινήσει ιδιαίτερα στη Γαλλία και αργότερα θα αξιολογήσουμε ε, τον αντίκτυπο του στους στόχους ε, της ε, βιώσιμης ανάπτυξης ε, και σε λίγους μήνες θα εξελίξουμε το τι θα κάνουμε στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Ευχαριστώ το ΕΛΚ για αυτό το οποίο ζήτησαν ιδίω όσον αφορά για την εξαναγκαστική εργασία των ανηλίκων κλπ. Διότι με ενδιαφέρουσες αυτές οι προτάσεις δεν μπορώ να συμφωνήσω ότι όταν συζητούμε για εμπόριο θα πρέπει να περιοριστούμε στην προβληματική για το τι γίνεται με τις επενδύσεις, για τις εμπορικές ροές κλπ. Νομίζω ότι η στρατηγική της Κομισιόν είναι ξεκάθαρη. Όταν λέμε εμπόριο για όλους εννοούμε την αύξηση των ορών, αλλά όμως υπάρχει και το θέμα της ε, αιτίας, το πώς μπορεί να γίνει ε, ε, μόχλευση ούτως με το ε, εμπόριο υπέρ των ε, ανθρώπων και οπότε ορθώς όλα αυτά τα θέματα τα συζητά και τα θέτει όσο ερωτήματα η Επιτροπή μας. Άκουσα όλα αυτά που λένε, άκουσα τι, που, που διαφέρουμε, άκουσα ποιος θέλει υποχρεωτικότητα ή όχι, είπαμε για τα μέταλλα, τα ορυκτά τέλο πάντων των σειράξεων και θα πρέπει να δούμε κατά πόσον ε, θα υπάρχει υπολογισμός υποχρεωτικών μέσων εάν η υπόθεση αυτή καλύψει και τις μικρομεζές επιχειρήσεις. Επίσης, σήμερα, νομίζω ότι υπάρχουν δύο προβλήματα όσον αφορά την εύρυθμη λειτουργία του εμπορίου. Πρώτα-πρώτα είναι ο θύμητο ανταγωνισμό. Όταν υπάρχει τέτοιο ανταγωνισμό που είναι οργανωμένο, αυτό είναι πολύ βλαπτικό για το εμπόριο, το διεθνέ εμπόριο. Επίση, ε, δεύτερο κουσούρι είναι ο προστατευτισμό. Άρα ε, το θέμα δεν είναι αν αυτά που λέμε πάνε προ την, την άλλη κατεύθυνση. Θα πρέπει ταυτόχρονα να καταπολεμήσουμε και τον θεμητό ανταγωνισμό και τον προστατευτισμό. Άρα με αυτό το κείμενο νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε αυτή την διπλή προσέγγιση και αυτό ήταν και το πνεύμα που διέπει το κείμενο το οποίο συντάξαμε. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Οπότε θα τα δούμε στις 30 Μαΐου και θα ψηφίσουμε στην Ίντα τον Ιούλιο. Και τώρα θα ξεκινήσει η συνεδρίαση των συντονιστών. Θα γίνει και κλεισμένο των θυρών, οπότε παρακαλώ όλοι που δεν είναι συντονιστές να αποχωρήσουν.